περασμένη εβδομάδα στην Τουρκία και πάλι έγινε ένα σεισμός. Πολλά άτομα και πάλι έχασαν τη ζωή τους, περίπου 700 άτομα και, και υπήρξαν και υλικέ ζημιέ στην περιοχή που ήδη υπέστη πριν από τρει εβδομάδες ένα σεισμό οι σκέψεις μας είναι με τους ε, Τούρκους συναδέλφους μας. Επίσης είχαμε πλημμύρες ε, στην Ιταλία και Νότια Γαλλία όπου έχασαν τη ζωή τους άνθρωποι και όπου εκεί υπήρχαν σημαντικές υλικές ζήμιες. Θα θέλαμε να συγχαρούμε ε, τις ομάδες διάσωσης ε, και τις διάφορες ε, τοπικές ομάδες που προσπάθησαν να βοηθήσουν αυτούς που επλήγησαν από τις θεομηνίες μας. Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους σε αυτές τις θεομηνίες και θα θέλαμε να εκφράσουμε και τις συμπάθειές μας σε αυτούς που παρέμειναν άστεγοι. Τις τελευταίες εβδομάδες. Την περασμένη εβδομάδα επισκέφθηκα την Λιβύη και την Τινησία Μιλήσαμε για την δημοκρατία και την οικονομία της αγοράς. Συζητήσαμε αυτά τα θέματα εκεί. Θέλουν να μάθουν από εμά πώς μπορούν να οικοδομήσουν δημοκρατικούς θεσμούς και πώς οι θεσμοί αυτοί είναι διαρθρωμένοι. Δεν μπορούμε βεβαίως να επιβάλλουμε τις ιδέες μας στους άλλους, αλλά νομίζω ότι οι Λίβοι ενδιαφέρθηκαν πάρα πολύ να μάθουν τα όσα είχαν να πω. Στην Τινησία συνήντησα τον Πρωθυπουργό, τον επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας και τους επικεφαλής των τεσσάρων ε, κυριωτέρων κομμάτων. Η Τινησία είναι ανοιχτή απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο λαός της ε, Τινησίας ε, δήλωσε ότι δεν έχει καμιά άλλη επιλογή από το να στραφεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για να την πάρει ως παράδειγμα. Μιλήσαμε για το θέμα του κράτους δικαίου και την ιδέα μιας κοινωνίας που θα περιλαμβάνει τους πάντες και θα επιτρέψει σε όλους να συμμετέχουν στην δημόσια ζωή ακόμη και στις γυναίκες η ε, ισότητα των ευκαιριών σε μια ανοιχτή κοινωνία για το θέμα αυτό. Τα τέσσερα βασικά κόμματα που κέρδισαν τις εκλογές είναι πρόθυμα να δημιουργήσουν μια δημοκρατική την Ισία και να συνεργαστούν με τους Ευρωπαίους. Επίσης, πέρασα περίπου μια εβδομάδα στα Δυτικά Βαλκάνια. Πήγα στην Κροατία, η οποία θα προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επισκέφθηκα τη Σερβία η οποία αντιμετωπίζει την πρόκληση της ομαλοποίησης των σχέσεων με το Κωσυφοπαίδιο ε, και που εφαρμόζει μια διαδικασία μεταρρυθμίσεων. Επισκέφθηκα την Βοσνία Ερζεγοβίνη που ε, προσπαθεί ε, να βγει από το αδιέξοδο το εσωτερικό. Επισκέφθηκα τη Σρεμπρενίτσα όπου εξ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέθεσα ένα ένα στεφάνι. Επίσης εκφράσαμε την συμπάθεια των μελών αυτού του Κοινοβουλίου προς τις οικογένειες των θυμάτων. Νομίζω ότι η Σρεμπρένιτσα είναι ένας σημαντικός τόπος προσκυνήματος, είναι πάρα πολύ σημαντικός για μας και πρέπει και εμείς να πηγαίνουμε εκεί για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε η διεσόμαση ε, ε, ποια είναι τα τρομερά πράγματα που μπορούν να συμβούν την Τετάρτη θα έχουμε μια σημαντική συζήτηση και θα έρθει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Βαν Ρομπόι, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μπαρόσο θα είναι παρόν και ο πρόεδρος του Eurogroup και πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Juncker θα είναι παρόν και θα έχουμε μια σημαντική συζήτηση και θα ήθελα όλα τα μέλη να ε, είναι παρόντα σε αυτή τη συζήτηση. Στις 2 σήμερα το απόγευμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Εφήβων ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Μεσογειακό έκλεισε τις συζητήσεις του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φιλοξένησε νέους από 40 χώρες που ε, κατανεμήθηκαν σε πέντε ομάδες εργασίας, κοινωνικός διάλογος, μετανάστευση και ενσωμάτωση, ισότητα ευκαιριών, ε, περιβάλλον, μεταφορές και ανανεώσιμες ενέργειες και η ανεργία και η απασχόληση. Ασχολήθηκαν με όλο αυτό το φάσμα των θεμάτων με το οποίο ασχολούμαστε και εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. η κοινωνία των πολιτών, ο κοινωνικός διάλογος, πραγματική ισότητα, πρόσβαση στην παιδεία, η εργασία και η προστασία του περιβάλλοντος. Η βαθμία ανάπτυξη μια ευήμερης κοινωνίας. Αυτά ήταν τα θέματα. Μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για τους νέους οι οποίοι βρέθηκαν εδώ, 250 νέοι από την περιοχή της Μεσογείου. Μερικοί από αυτούς είναι ακόμα εδώ, εδώ πάνω στα θεωρία. Εκεί που κάθεστε σήμερα αξιότιμα μέλη καθόντουσαν πριν από μερικές μέρες αυτοί οι νέοι, αυτοί οι έφηβοι. Θα ήθελα να καλέσω τα μέλη να συμμετάσχουν σε μια διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 23 Νοεμβρίου υψηλού επίπεδου για τα ανθρώπινα δικαιώματα όπου θα φιλοξενήσουμε επίσης ε, αυτούς ε, που του βραβείου Σαχάροφ, 12 από αυτούς ε, επιβεβαίωσαν την παρουσία τους. Βεβαίως όλοι δεν θα μπορέσουν να έρθουν, αλλά νομίζω ότι πάρα πολλοί από αυτούς θα ήθελαν να έρθουν στη διάσκεψη αυτή. Θα υπάρξει μια ευρεία συζήτηση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους υπερεσπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η διάσκεψη αυτή θα λάβει χώρα στις 23 Νοεμβρίου στο τέλος της ημέρας θα έχουμε μια ανοιχτή συνάντηση στο Beaux-Arts με πολίτες των Βρυξελών. Και τέλος, μερικά λυπηρές ειδήσει, λυπηρό νέο για το θάνατο του Willy de Klerk. Χάσαμε έναν Ευρωπαίο ε, και Βέλγο ηγέτη ο οποίος ήταν για πάνω από 25 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν επικεφαλής της ομάδας των φιλελευθέρων και ήταν σε μια από τις μόνιμες επιτροπές πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήταν επίσης επίτροπος και ε, υπήρξε αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως του Βελγίου. Θα ήθελα να σηκωθείτε αξιότιμα μέλη και να τηρήσετε ενός λεπτού σιγή. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα